Έχουν παρατηρήσεις. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Ας περάσουμε στις ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 211 του κανονισμού, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προτείνει την εξή ερμηνεία του άρθρου 187 όσον αφορά τη σύνθεση των επιτροπών και των αναπληρωτικών μελών. Σε περίπτωση ε, θέση ένα αναπληρωματικό μέλος ορίζεται από την ίδια πολιτική ομάδα ε, σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 5 ή αν δεν υπάρχει τέτοια προσωρινή αντικατάσταση μέχρι τον διορισμό νέου μέλους ε, πλήρους μέλους. Ε, αυτό βασίζεται σε απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με την αριθμητική σύνθεση της Επιτροπής και αποσκοπεί στην εξασφάλιση κατά την ψηφοφορία ικανού αριθμού ε, εκπροσώπων των ε, πολιτικών ε, ομάδων σε σχέση με την καινή αυτή θέση. Αυτό ισχύει σε, εκτός από την περίπτωση που μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 προβουλευτές αντιτίθεται πριν από την άνοιξη της επόμενης συνόδου. Το κείμενο της ερμηνείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ε, Seance on Direct. Δεύτερη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Λιθουανίας κοινοποίησαν στο Κοινοβούλιο την ε, εκλογή της συναδέλφου Τζουστίνα Βίτκα Ουσκάιτε ε, ως αντικαταστάτρια του κυρίου Βίκτορ Ουσπάσκης ε, με ισχύ από 21 Νοεμβρίου 2012. Οι αρμόδιες αρχές